ευχαριστώ. Καλή μέρα των γυναικών. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Παίρνουμε και τι παρεμβάσει διάρκεια ενός λεπτού. May I remind you it's one minute speech, so please the time. Παρακαλώ να μιλάτε για ένα λεπτό. Η κυρία Μπόκτσορ είναι η πρώτη που παίρνει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και θα ήθελα να τονίσω ότι στις 28 Φεβρουαρίου η Ακαδημία η Αμερικανική έδωσε το Όσκαρ, μίλησε τα Όσκαρ. Μετά από 40 χρόνια μας ήταν ενθουσιασμένοι για την τελετή διότι είχαμε υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερη ταινία. Ο γιο του Σαούλ, του κυρίου Γέλε, του Λάσλο Γέλε, κέρδισε το αγαλματίδιο αυτό και έφερε την επιτυχία και στην Ουγγαρία και στην Ευρώπη. Κέρδισε πολλά βραβεία στο Φεστιβάλ των Κανών. Έχει πάρει τη Χρυσή Σφαίρα και, και το βραβείο ανεξαρτήτου πνεύματος πήρε αργότερα, μια εβδομάδα μετά το Όσκαρ αρκετές επιτυχίες είχαμε και πριν αυτή την ταινία τα τελευταία χρόνια και όλα αυτά εμπλουτίζουν τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό. Είναι πολύ σημαντικό να ε, στηρίζουμε την ευρωπαϊκή δημιουργία και αυτό είναι επιτυχία για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο όπως είναι και για την Ουγγαρία. Εξίσου σημαντικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Καπασαλουρίς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πατήτης είναι μια μολυσματική ασθένεια που 14 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από αυτήν και βλέπουμε ότι ένα μικρό ποσοστό είναι εκείνο το οποίο είναι γνωστό για τους όσους έχουν μολυνθεί και υπάρχει κίνδυνος της μετάδοσης ε, ε, ε, μέσω του αίματος, μετάγγισης και εδώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διότι η μολυσματική αυτή ασθένεια οδηγεί σε κύρωση του ύπατος ή σε περιπτώσεις καρκίνων. Αυτή τη στιγμή πρωτόκολλος ευρωπαϊκό επίπεδο που λειτουργεί, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανείχνευση και με την ε, ε, συντονισμένη δράση κρατών μελών για τη δημιουργία ενός μητρώου. Και όπως ε, γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν καινοτόμα φάρμακα που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την περίπτωση αυτή τη ασθένεια. Είναι όμω μεγάλη η πρόκληση για τα υγειονομικά συστήματα όπω τη Ισπανία για παράδειγμα που υφίστανται μεγάλε περικοπέ και πιέσει. Ε, μπορεί να εκκρίζωθεί αυτή η μολυσματική ασθένεια και αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει, να καταρτήσει ένα πρόγραμμα για την εκκρίζωση αυτή τη ασθένεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πρέτσελ το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την Ολομέλεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο άμεσο προσεχές διάστημα θα ασχοληθούμε περισσότερο και με το σκάνδαλο όπως αποκαλείται Volkswagen και δημιουργήσαμε, καταρτήσαμε και μια επιτροπή γι' αυτό. Τα σκάνδαλα της Volkswagen όπως αποκαλούνται η υπόθεση όμως αυτή είναι πιο περίπλοκη από αυτό τον χαρακτηρισμό, αυτό τον τίτλο. Το Διεθνές Συμβούλιο για τις Καθαρές Μεταφορές, ICCT, όπως αφορά τις ΙΠΑ και τις υπηρεσίες που απεκάλυψαν αυτά τα κακό κείμενα, σε πολλές δοκιμασίες απέρευσε το συμπέρασμα ότι υπάρχουν και προβλήματα και με άλλους αυτοκινήτων, ιδιαίτερα Citroën, Opel και Fiat Δύο από αυτούς, η Opel και η Fiat, ανήκουν σε αμερικανικές αυτοβιομηχανίες ως επιχειρήσεις. Και γι' αυτό θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας σε αυτό το θέμα για να αναγνωρίσετε και να δείτε ότι πρόκειται για κάτι παραπάνω από την εμπλοκή μόνο μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπάρχει οικονομικός πόλεμος εδώ που έχει ξεσπάσει από συμφέροντα βιομηχανιών της των ΗΠΑ έναντι ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Κυρία Σήμερα ένα email από την Κάρμ Λαγκάρ που είναι καθηγήτρια από το West Cork στην Ιρλανδία. Η Κάρμεν είναι θελόντρια στη Λέρο και βοηθάει τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες κρατούνται σε κέντρα που δεν έχουν επαρκή διατροφή και αποχέτευση. Εθελοντικέ οργανώσει ήδη έχουν υπερφορτωθεί και προσπαθούν να βοηθήσουν όμω. Η Κάρμελ έχει συγκλονιστεί και οι πιο βασικέ ανάγκε των προσφύγων, τρόφιμα και νερό, η υγεία δεν καλύπτονται. Και έγραψε σε όλου του Ιρλανδού Ευρωβουλευτέ ζητώντα βοήθεια. Ήλπιζα ότι το σημερινό Συμβούλιο θα έδινε κάποια λύση, κάποιο πλαίσιο, κάποια ελπίδα. Αλλά για μία ακόμη φορά τι είδαμε, κανένα, καμία λύση, κανένα ψήφισμα, τίποτα. Απογοητεύομαι. Και Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε 130.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα. Μόνο φέτος. Μόνο συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορεί να αρχίσει να λύνει το πρόβλημα. Αν οι ηγέτες μας δεν μπορούν να πλησιώσουν μια λύση, όσο και δύσκολο και αν είναι αυτό, όχι μόνο θα υποφέρουν οι μετανάστες, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφέρει. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίλβα Ροντρίγκε. Σένρα Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στο πρωτογενή τομέα είναι το αίτιο των πάνδυνων που υφίστανται στη δική μου χώρα οι πολίτες. Έχουμε ποσοστώσεις και τον νόμο για τη Γαλλικία, για τη Γεωργία και την ετικετοποίηση όσον αφορά τις κονσέρβες αλλιευμάτων ψαριών και για το, τη γεωργική παραγωγή και τις αγορές γεωργικών προϊόντων όπως συμβαίνει για τα γαλακτοκομικά χαμηλές τιμές των γεωργικών προϊόντων που είναι μια σωστή και καλή απόδειξη της μεγάλης κρίσης που διανύουμε στον γεωργικό και αλλιευτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να αντιδράσει. Πρέπει να αλλάξει η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή αλλιευτική πολιτική για να διασφαλιστεί το μέσο διαβίωσης χιλιάδων, μυριάδων πολιτών στη Γαλλικία και στο νότο της Ευρώπης. Δεν θα υπάρξει μέλλον για την Ευρώπη αν αυτές οι πολιτικές εξόντωσης των λαών και των πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαραγκάλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ σήμερα για άλλη μία φορά. Έχουμε τη συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για τους πρόσφυγες αν αυτές οι συζητήσεις και διαβουλεύσεις δεν λάβουν υπόψη ε, συγκεκριμένα ζητήματα που είναι κατεπήγοντα δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε καμιά νέα συμφωνία. Έχουμε και τις πολιτικές ε, της ε, Τουρκίας για το ΠΚΚ. Μπορεί κανείς ίσως να μην βλέπει τα όσα συμβαίνουν στον Διαρμπακύρ και στην περιοχή των Κούρδων στο Κουρδιστάν. Οι οποίοι Κούρδοι βρίσκονται σε, σε μια πολιορκία. Μπορεί η Ευρώπη να αγνοεί τις συλλήψεις δικηγόρων και την δίωξη πολιτών. Μπορεί η Ευρώπη να είναι αδιάφορη για τους πρόσφυγες και όσους πνίγονται στις ακτές της Λέσβου. Μπορεί κανείς ε, σε σχέση με τον αποκλεισμό των Βαλκανίων ε, η Ευρώπη να δεχθεί τα όσα συμβαίνουν. Έχουμε εδώ την, ε, την τιμωρία που υφίσταται ένα κράτος μέλος η Ελλάδα για όσους μπορούν και εισέρχονται σε αυτή τη χώρα αλλά δεν μπορούν να εξέλθουν από αυτήν. Πρέπει εδώ η Ευρώπη επιτέλους να τα δει και να δράσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Άκερ έχει το λόγο. Θα ήθελα να φέρω ένα θέμα εκλογικής περιφέρειας και να πω ότι είμαι κάθετα αντίθετος με την πρόταση της νέας διελεύσεως του ε, Τάμεσης, το Θόρεκ. Δεν λέω αν είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κακή. Το Θόροκ. Αυτή η νέα γέφυρα θα αυξήσει την διέλευση, θα αυξήσει την μόλυνση, θα αυξήσει τη συμφόρηση ε, στο δικό δίκτυο και θα αφαιρέσει και σπίτι από τους κατοίκους. Αυτή η κυβέρνηση ε, θέλουν να ρίξουν στο θόρο αυτή τη λύση. Η συντηρητική. Η κυβέρνηση μπορεί να με την εκλογική περιφέρεια, αλλά ε, τελικά στη χειρότερη θέση καταλήξει η κυβέρνηση. Θόροκ δεν είναι μόνο η δική μου εκλογική περιφέρεια, είναι το σπίτι μου. Και μαζί ενωμένοι θα πολεμήσουμε αυτή την διέλευση ε, σε όλο τη... μέχρι τέλους. Thank you. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπίλντε έχει το λόγο τώρα. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 800 φάλαινες σφαγιάζονται κάθε χρόνο στις Φερόες νήσους με μεγάλη διαφορία που επικρατεί Πρόκειται περισσότερε φανέ που σκοτώνται από ό,τι χρειάζεται για την κατανάλωση του τοπικού πληθυσμού. Και έτσι περαιτέρω η κατανάλωση του κρέατο τη φάλαινα δημιουργεί κίνδυνο για τη υγεία του ανθρώπου, διότι υπάρχει υδράργυρο και τοξίνε. Τα παιδιά ακόμα μπορούν να βλέπουν τη θανάτωση και τον τεμαχισμό των φαλενών. Ακόμα και αν είναι οι είναι αυτόνομες νομικώς από την Δανία και αν σέβομαι πάρα πολύ τι παραδόσεις και τι ανάγκε τη διατροφή, όμω είναι κατεπίγουσα ανάγκη να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει με τι αρχέ των νησών Φερόε και με τη Δανία για να ρυθμιστεί αυτό το θέμα και να διαπραγματευτεί κάθε κίνδυνο για την υγεία και να σταματήσει σταδιακά αυτή η πρακτική η οποία είναι πολύ κακή. Λοιπόν, μπορούμε να κρίνουμε τον πολιτισμό ενό λαού με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα ζώα. Είναι και, η ώρα να αντιδράσουμε και να σταματήσουμε να στηρίζουμε με την σιωπή μα ε, αυτή την σφαγή. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Μάτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένας έφηβος στο Καράκασα απεβίωσε αναμένοντας φάρμακα που μπορούσαν να τον είχαν διασώσει. Είναι φοβερό το ότι δεν γνωρίζουμε για παρόμοιες περιπτώσεις. Η κατάσταση των κατοίκων της Βενεζουέλας όπου η πρόσβαση σε φάρμακα δημιουργεί τέτοιες δραματικές καταστάσεις έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση και δεν μπορούμε να είμαστε απαθείς ε, ενώπιον αυτής της ε, κρίσης. Ε, ούτε αξίζουν τα άτομα αυτά οι πολίτες της Βενεζουέλας να υφίστανται αυτή την κατάσταση και να βρίσκονται στις φυλακές Αντώνιο Λόπες, Λεντέσμα και άλλοι που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση από τον προηγούμενο Αύγουστο. Όλοι αυτοί είναι πραγματικά πολιτικοί κρατούμενοι και γι' αυτό είναι έσχος ότι υπάρχουν κάποια άτομα στην Ολομέλεια που δεν αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα για το ότι δηλαδή πρέπει να θεωρούνται πολιτικοί κρατούμενοι ως ε, και την ε, ε, απελευθέρωση κάποιων την ορτάζουν ως απελευθέρωση και δικαίωση κάποιου ενώ ήταν τρομοκράτης της ΕΤΑ. Για τους και τους ε, φίλους τους ε, ε, βλέπουμε με τη μεγαλύτερη περιφρόνηση αυτή την στάση τους. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εδώ και χρόνια η παραγωγή των ε, αποβλήτων ε, που κοστίζει τεράστια ποσά και όλα με την επιβάρηση του περιβάλλοντος όταν αυτά καταλήγουν στη θάλασσα. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι υφίστανται τα πάνδυνα εδώ οι πολίτες. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω για το πρόβλημα των ε, αποβλήτων στην ακτή της Κροατίας. Βλέπουμε ότι εδώ επιβαρύνονται ακτές της Κροατίας και ομόρων χωρών. Βλέπουμε εδώ ότι όπως το Σερτενίκ αρχές και επιχειρήσεις οδηγούν, ε, ανέχονται αυτή την κατάσταση. Αυτά τα απόβλητα έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις ε, διότι οι καθαρές ακτές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Κροατία και πρέπει εδώ να δούμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εργαστούμε και να συνεργαστούμε για να διασφαλιστεί μέχρι το 2020 η καλή ποιότητα του ε, συστήματος ε, του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κυρία Να σας επιστήσω την προσοχή σε κάτι. Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα νομοθετούν και θα πρέπει να έχουν σαφείς κανόνες που θεσπίζουν και κανονισμούς. Γιατί καμιά φορά η ευρωπαϊκή νομοθεσία εμποδίζει διάφορους φορεί από το να μπορούν να λειτουργούν σωστά και αποτελεσματικά. Αυτό είναι και επιβλαβές όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι σημαντικά όλα αυτά ε, βλέποντα την αναθωρημένη οδηγία για την μετάθεση, την απόσπαση των εργαζομένων. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λησμόνησε ότι η εφαρμοστική οδηγία 2014 είναι αυτή που υλοποιείται και διάφορα κράτη-μέλη και διάφοροι φορείς ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην θεσπίσει νέα νομοθεσία. Και η αναθεώρηση ε, της νομοθεσίας θα λάβει χώρα ανεξάρτητα από τις εφαρμοστικές διατάξεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκραπίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί. Η παγκοσμιοποίηση ε, ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να παραμένει μόνο ένα σύνθημα. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την πρόσβασή του σε αγορέ τρίτων χωρών και να την εγγυηθούμε. 90% τη ανάπτυξη θα προέρχεται από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμούν οι ειδικοί και το 60% της ανάπτυξης θα είναι από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό φέρει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δομολογήσει αυτή τη διαδικασία υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διεθνοποίησης της δραστηριότητάς τους. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται την συμφωνία TTIP και την διμερή συμφωνία με την Κίνα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ε, πρόσβασης ε, των επιχειρήσεων σε αυτές τις αγορές να ε, βοηθήσει τις επιχειρήσεις για τη διεθνοποίηση της δραστηριότητάς τους θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι ισότιμη όρια ανταγωνισμού ακόμη και σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητες δυσκολίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός Ένωσης αγοράς. Ευχαριστούμε κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα σήμερα να κάνω την μονόλεπτη ομιλία μου για την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, και, και Καλνιέτη, θα ήθελα να τους συγχαρώ για την πρόταση που υπέβαλαν. Είναι λογική και πρέπει να εξασφαλίσουμε όντως την παροχή του φυσικού αερίου και μετά από την COP21 θα πρέπει να φροντίσουμε να καλύψουμε και την αυξημένη ανάγκη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τι είναι φεδρική λύση. Ποια είναι αυτή το φυσικό αέριο με το υγροποιημένο φυσικό αερίο και κυρίως αυτά που συμβαίνουν στη ΣΥΠΑ, στην Αυστραλία και στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα λογικές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τερματική σταθμή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, όπως και στη δική μου εκλογική περιφέρεια, νομίζω ότι σε τοπικό επίπεδο ε, θα μας βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε και το φυσικό αέριο που έρχεται από τη ΣΥΠΑ, γιατί είμαστε ο κοντινότερος λιμένας ε, μετά τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Επίσης ε, ελπίζουμε να ε, αναπτυχθούν αυτή η τερματική σταθμή στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε κυρία Ward. Ευχαριστώ. Να επιστήσω την προσοχή στην πολύ κακή ανθρωπιστική κατάσταση που κρατεί τις πρόσφυγες που ζουν σε φρικτές συνθήκες, σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στα σύνορά μας εκτίθενται στα στοιχεία τα καιρικά και οι πρόσφυγες όπως είναι στο Καλέ και στη Δουνκέρκη, στις ζούγκλες εκεί είδαν ότι πλημμύρισαν τα, οι καταβλισμοί τους και έτυχαν πολύ περιορισμένες υποστήριξη για να περάσουν το χειμώνα. Τα βάσανά τους αντιβαίνουν τις βασικές προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια. Πάνω σε αυτές τις αρχές έχει δοθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα παιδιά και γυναίκες στα στατόπεδα αυτά δεν έχουν τις βασικές ανάγκες τους καλυπτόμενες. Η υγεία, παιδεία, και υγειονομική περίθαλψη. Δεν τους βοηθούμε εμείς, αλλά μπαίνουν οι διακινητές. Αντί να υπάρχει ανθρωπιστική απάντηση, είδαμε βία της αστυνομίας και επιθετικότητα ε, και εκδιώχθηκαν βία. Είναι τραγικό εκείνοι που έπρεπε να ξεφύγουν από τον Ντάι στη Συρία, από τη Φρίκη και να κινδυνεύσουν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να βρουν καταφύγιο, τώρα αντιμετωπίζουν τέτοια φρικτή ε, αντιμετώπιση από τους συντρόφους μας τους Ευρωπαίους. Εμείς που λαμβάνουμε τις αποφάσεις θα πρέπει να δούμε με τα μάτια μας αυτούς τους καταβλισμούς και να μιλήσουμε με κάποιες πρόσφυγες, εμείς οι ίδιοι, όπως έκανα και εγώ. Και Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην σημερινή οικονομική συγκυρία τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά θεσμικά οργανά πρέπει να δράσουν αποτελεσματικά και να συντονίζονται μεταξύ τους. Κάνω λόγο για την παραγωγή διότι έχουμε, ε, ε έχουμε έλλειμμα 300.000 τόνων όσον αφορά την παραγωγή πρόβειου κρέατος και βλέπουμε ότι αυτή η ανάγκη δεν καλύπτεται. Γι' αυτό χρειαζόμαστε φιλόδοξα σχέδια για να, μπορέσουν, να, να μπορέσει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα του πρόβειου κρέατος και της εκτροφής προβάτων ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπάρχει τέτοιο έλλειμμα όπως η τη Ρουμανία που έχει το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης για τον τομέα τομέα του πρόβειου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να απευθύνω έκκληση να βελτιωθεί η κατάσταση της Ρουμανίας και να βοηθηθεί η Ρουμανία από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να βελτιωθεί το δυναμικό της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Uh, η κυρία Βον Στόρκ έχει το λόγο. Μάλιστα σήμερα συνήλθαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης και της Τουρκίας για την προσφυγική κρίση για τα Βαλκάνια ε, που υπάρχει η πρόθεση να κλείσει ο διάβλος των ε, δυνατοτήτων ε, πρόσβασης των προσφύγων μέσω των Βαλκανίων. Δεν έχει όμως κάποιο ενδιαφέρον ή συμφέρον η Ευρωπαϊκή ή η Τουρκία να παραμείνει ανοιχτή αυτή διάβλος διότι τότε δεν μπορεί να πιέσει, να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι ε, σήμερα δεν ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προβλήματα τα οποία εφίστανται στην Τουρκία όπως το ότι κλείνει εφημερίδα και διώκονται δημοσιογράφοι. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να αποτελεί την λύση του προβλήματος. Επικρίσεις εις βάρος της Τουρκίας εκεί όπου είναι αναγκαίο, ναι. Ωστόσο το να βασιστούμε στην Τουρκία για να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση, όχι. Να μην το κάνουμε. Ευχαριστώ ο κύριος Βιέγκας. As leis do mercado, οι νόμοι της αγοράς, η ευμεταβλητότητα των τιμών των γεωργικών προϊόντων υπονομεύουν τις ε, γεωργικές δραστηριότητες που η εμβέλειά τους ξεπερνά κατά πολύ την πραγματική τους διάσταση απλά οικονομική. Βλέπουμε ότι κλείνουν επιχειρήσεις και πρέπει άμεσα να λάβουμε μέτρα και να βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε τις ε, δυνάμεις της αγοράς ε, ώστε να δράσουν αποτελεσματικά. Και πρέπει εδώ να υπάρξουν και οι δράσει ώστε να μπορούν να διασφαλίζονται οι τιμέ των προϊόντων τους. Φτάνει πια με τις απάτες ει βάρος ε, των γεωργών σε σχέση με κάποια εικονικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η κατάστασή του παρόλη την λήψη αυτών των μέτρων μόνο η δημόσια βελτίωση της προσφοράς ε, όσον αφορά και την δυνατότητα ζήτησης μπορεί να δώσει μια εφορία όσον αφορά τον κοινωνικό περιβαλλοντικό τομέα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τόμς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ οι δείκτες, οι στατιστικοί δείκτες όσον αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Σλοβενία είναι καλύτεροι, έχουν βελτιωθεί. Αυτό είναι πολύ καλό βέβαια. Ωστόσο δεν το ζουν και το βιώνουν αυτό με τη βελτίωση των δικτών οι Σλοβαίνοι στη ζωή τους. Διότι τα προβλήματα των πολιτών εξακολουθούν και υφίστανται στη χώρα μας. Πρέπει να μεταρρυθμιστούν τα συστήματα της ε, ε, περίθαλψης, της υγείας, ε, να υπάρξει βελτίωση όσον αφορά τη φορολογία επιχειρήσεων. Πρέπει να αλλάξει επίσης και το νομικό πλαίσιο και όσον αφορά και τις ιδιωτικοποιήσεις. Ναι, μεν εφαρμόζεται η τάση των ιδιωτικοποιήσεων αλλά όχι στο αναγκαίο μέτρο. Και για τις τράπεζες επίσης έχουμε και την κρίση των προσφύγων, την προσφυγική κρίση που δεν μπορεί να είναι πρόσχημα για να τερματιστούν και να πάψουν οι μεταρρυθμίσεις. Τα μία τώρα, τα δημόσια μία, όσον αφορά τη διαχείρισή τους. Παρουσιάζουν προβλήματα δομών και διαθρώσεων. Γι' αυτό ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση στη Σλοβενία, τη χώρα μου. Ευχαριστώ κ. Μπράνεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά για τους γεωργούς της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου όταν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Άγκρη Union που είναι συμβουλευτική επιχείρηση στην Βρετανία, μόνο 10% από τις εκμεταλλεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα επιβίωναν σήμερα άμα σταματήσουν οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει κάποιο χώρο Θα συμβεί αν τελικά αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι επιδοτήσει δίνουν 50 με 60% ε, των εισοδημάτων των εγκαταλέψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, αν φύγουμε τελικά θα είναι άλμα στο σκοτάδι, ένα ταξίδι αχαρτογράφητο. Από πλευρά των γεωργών όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφορά μόνο την κοινή αγροτική πολιτική. Οι γεωργοί μα έχουν και τα ωφέλη του εμπορίου και τη ελεύθερη ροή των εργαζομένων. Η γεωργία μα εξαρτάται πολύ από πρόσβαση στην ενιαία αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πουλήσει τα προϊόντα. Περίπου δύο τρίτα τη γεωργικών εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παραγωγοί μα ενδεχομένω θα αντιμετωπίσουν δασμού από 11 μέχρι 48% ε, για να μπουν στην ενιαία αγορά. Θα πρέπει οι γεωργοί να ψηφίσουν να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς η προσφυγική κρίση στην ελλάδα έχει πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις καθώς οι πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί μέχρι στιγμής ανέρχονται σε σαράντα και ο αριθμός τους θα αυξηθεί επιπλέον κατά εκατό στο τέλος του μηνός. η τουρκία συνεχίζει να υποθάλπει τα δουλεμπορικά κυκλώματα μεταφοράς προσφύγων στα νησιά του αιγαίου και η μετεγκατάσταση έχει μείνει στα χαρτιά αφού από τους 60.400 πρόσφυγες έχουν αναχωρήσει από την ελλάδα λιγότεροι από 400 η ευρωπαϊκή ένωση με την πολιτική της έχει μετατρέψει την ελλάδα σε ένα απέραντο προσφυγικό ταχάου. μόνη λύση να στηριχτεί πλέον ο ελληνικός λαός στις δικές του δυνάμεις. η ελλάδα λοιπόν πρέπει να αποχωρήσει από τη σέγγεν για να πάψει έτσι να αποτελεί μαγνήτη για τους πρόσφυγες που έρχονται στην πατρίδα μου αντί να πάνε στη βουλγαρία γιατί η ελλάδα ως χώρα σέγγεν χορηγεί στους πρόσφυγες ταξιδιωτικά έγγραφα τύπου σέγγεν που τους επιτρέπουν να φτάσουν στη γερμανία επιπλέον η ελλάδα πρέπει να αναστείλει το δουβλίνο τρία να επιβάλει οικονομικό εμπάργκο στα σκόπια και την αλβανία ως αντίπεινα προκειμένου να αναγκάσει τις χώρες αυτές να ανοίξουν για τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες τα σύνορά τους τα οποία έχουν κλείσει παράνομα όπως δήλωσε και ο γενικός γραμματέας του οηε κύριος μπαν κι ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόγκορ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. πολύ. Μπορεί ίσω να είναι μια έκπληξη την οποία δυστυχώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να βιώσουμε αυτή. Είχαμε μια εκδήλωση για τι μειονότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να επιστήσω την προσοχή σα ότι σε αυτή την εκδήλωση ε, δεν υπήρξε η αποκατάσταση του δικαίου. Δηλαδή τι συνέβη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια άτομα προσπάθησαν να εκφράσουν τις απόψεις τους με τρόπο απαράδεκτο, με ιδιαίτερα επιθετικό κιόλα. και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Όλα αυτά στη συνθήκη καθορίζονται. Ποιοι είναι οι όροι και προϋποθέσεις και οι αξίες στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο αλληλοσεβασμός και ο σεβασμός των απόψεων των άλλων της διαφορετικότητας. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, ως θεματοφύλακα των συνθήκων να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην ενδιαφέρεται μόνο για οικονομικά προβλήματα αλλά και για άλλα ζητήματα και προβλήματα. Η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία της άποψης είναι πολύ, ε, πολύ σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα έλεγα ότι η ίδια ιστορία, η ίδια ιστορία είναι κάτι το οποίο εξ, εξηγεί το τι συμβαίνει. Υπάρχουν πάντα κάποιοι οι οποίοι βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα και οι οποίοι φυστανε διακρίσεις και αρνητική μεταχείριση και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιβάλλουν το εννοούμενο δίκαιο από πλευράς τους και πολλές φορές ε, η δημοκρατία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω μιας τέτοιας Τέτοιου είδου άτομα πολλές φορές ε, οδηγούν ε, ίσως και σε καταστάσεις που όχι μόνο είναι προβληματικές αλλά και χαοτικές. Ο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας για παράδειγμα έκανε διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν δημοκρατικά ή δημοκρατικές πράξεις. Την τελευταία κιόλας εβδομάδα, πολύ πρόσφατα, ε, δικοί του ε, άνθρωποι ε, επομίστηκαν καθήκοντα εκτέλεσης ε, αρμοδιοτέ ότι θα πρέπει να διεξαχθεί λέει δημοψήφισμα για τα θέματα των προσφύγων. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει χαοτική κατάσταση λοιπόν στην Ουγγαρία. Μετά τη συζήτηση Ιανουαρίου για τους Βρετανούς και άλλους πολίτες που είναι φυλακισμένοι στην Ινδία, όπως και τον Νίκ Ντόν που στην εκλογική μου περιφέρεια, η, η αίτησή τους για απελευθέρωση δεν ε, έγινε δεκτή, ενώ περιμένουν να εκδικαστεί η έφεση. Λοιπόν, η εταιρεία θα έπρεπε να είναι υπεύθυνη και όχι τα άτομα ε, που δούλευαν για αυτούς, ε, που βρήθηκαν στη λάθος περιοχή, στη λάθος στιγμή. Είναι ε, προσωπικό ασφαλείας αυτοί οι άνθρωποι που προστάτευαν το κοινό και είδα και τα προσόντα τους. Έχω εδώ αντίγραφα των εξαγωγικών αδειών που έδειχνε ότι τα όπλα που εξήχθησαν εξήχθησαν νομίμως και εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων. Εγώ σέβομαι την ειδική κυβέρνηση που σταθεί να καταπολεμήσει τα παράνομα όπλα. Όμως σε αυτή την περίπτωση έπιασαν λάθος ανθρώπους. Καλό την ειδική κυβέρνηση κατεπηγόντω να αναθεωρήσει την υπόθεση και να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση ε, του ε, ανθρώπου αυτού που ανήκει στην εκλογική μου περιφέρεια. Ο κύριος Ζεντόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, η κατάσταση στα ελληνοσκοπιανά σύνορα ε, είναι αβάστακτοι, ανυπόφοροι. Η Ελλάδα δεν έχει αρχίσει ε, τους ε, ελέγχους όπως θα έπρεπε κατά την άφηξη των προσφύγων. Έτσι θα έπρεπε να γίνεται, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Γι' αυτό χιλιάδες άνθρωποι τώρα συνοστίζονται στα σύνορα προσπαθώντας να φτάσουν στην κεντρική Ευρώπη μέσα από αυτές τις χώρες διέλευσης. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως η μη κατάλληλη διαχείριση των συνόρων επιτρέπει σε επικίνδυνα άτομα να εισέρχονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να ανακόψουμε την ροή και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου όσου παραμένουν εδώ, συμπεριλαμβανομένων και των διερμηνέων. Ο κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, αναφέρω ότι για πολλές κοινότητες στη χώρα μου τα κοινωνικές, κοινωτικές επιδοτήσεις είναι μοναδική πηγή χρημάτων. Όμως ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές. Ε, θα πρέπει να ζητήσουμε από τη ρουμανική κυβέρνηση να αναλάβει κατεπηγόντως μέτρα ούτω ώστε η Ήπεθρος να έχει πρόσβαση άμεση στα κοινωτικά κονδύλια. Χρειαζόμαστε απλοποιημένες διαδικασίες και ένα συγκεκριμένο έντυπο που θα μπορούν να υποβάλουν ε, ταχύτατα. Μετά τις ε, τοπικές εκλογές ε, όλοι οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να εστιάζουν την προσπάθειά τους στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο ένα χρόνο από την κοινωνική χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε καλύτερη πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Ευχαριστούμε και ε, καλή ημέρα γυναικών. Ε, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες τις συναδέλφους. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Κάπελ, ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι βιομηχανίες έχουν επιπτώσεις στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρήπων ε, και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα τέλη είναι διπλάσια στις, ε, στην Ευρώπη σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και αφήστε που μειώθηκαν οι εκπομπές στη ΣΥΠΑ χωρίς το σύστημα δικαιωμάτων, ε, ε, ε, ε εμπορίας δικαιωμάτων ρήπων έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από εμά χωρίς κανένα τέτοιο σύστημα. Η Κίνα στη Χαλιβουργία έχει υπερβολική δυναμικότητα λόγω των κρατικών επιδοτήσεων και εμείς ε, υποφέρουμε από τα τέλη που πληρώνει η βιομηχανία και από αυτό το σύστημα ε, εμπορίας δικαιωμάτων. Έχουν επίσης για τη Χαλιβουργία επιβληθεί και οι κυρώσεις ε, και μέτρα αντι κατά της Κίνας αυτό όμως επηρεάζει μόνο κατά 40 έως 60% ε, της εξαγωγής της Κίνας. Μπορούμε να πούμε ότι τελικά ε, ο τομέας της χαλιβουργίας ε, θα πρέπει να συρρυχνωθεί. Κυρία Σακορά. Η αρχηγή των 28 μελών της Ευρώπης των 500 εκατομμυρίων συνεδριάζουν σήμερα πάνω στα συντρίμια της Ενωμένης ΕΕ. Κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και με τη σημερινή τη μορφή, δεν γίνεται να υπάρξει χωρίς τον σεβασμό στους κοινού αγώνες, στις κοινέ ευθύνε και στις κοινέ δεσμεύσεις. Είναι τουλάχιστον ηρωνία να συζητάμε για Ενωμένη Ευρώπη με κλειστά σύνορα, φτωχοποιημένους λαούς και χιλιάδες εξαθλιωμένου πρόσφυγες μονομερείς αποφάσεις ενάντια στις αρχές αλληλεγγύης και του καταμερισμού των ευθυνών που παίρνονται στο όνομα μικροπολιτικών συμφερόντων εθνικής κατανάλωσης το μόνο που καταφέρνουν είναι να γιγαντώνουν τη μυσαλλοδοξία και τα φασιστικά στοιχεία. οι κοινέ αποφάσει και δεσμεύσει δεν υλοποιούνται οι διεθνεί συνθήκε έχουν μετατραπεί σε κουρελόχαρτα και η ευρωπαϊκή επιτροπή περιορίζεται σε ευχολόγια. κύριοι συνάδελφοι κυρία πρόεδρε αλήθεια πιστεύετε ότι μπορεί η ελλάδα να σηκώσει την ευθύνη ολόκληρης της ευρώπης για το προσφυγικό; αλήθεια πιστεύετε ότι η λύση είναι τα οικονομικά ανταλλάγματα; η μόνη λύση είναι η ασφαλής δρόμη για τους πρόσφυγες και αναλογική φιλοξενία τους φυσικά από όλα τα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Thank you. Το κυνήγι λαγών με σκυλιά γκάλγο είναι μια παράδοση στην Ισπανία, όμω. Ε, ε, Πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι εκατομμύρια κυνήγοι ε, κάνουν αυτή τη βαρβαρότητα κακοποιώντας 50.000 ε, ε, ζώα κάθε χρόνο, τα κροτηριάζουν, τα καίνε ζωντανά, τα αφήνουν να πεθάνουν, λεπορούν, κακοποιούν αυτά τα ζώα, ορισμένοι χρησιμοποιούν και ένα σκηνή για να κρεμάσουν τα ζώα, ώστε να ασφικτιούν για όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα γίνεται. Ε, είναι ε, ε, πραγματικά νεκροταφεία ζωντανών ζώων ε, είναι απαράδεκτες αυτές οι πρακτικές ε, αντιτάσσονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το ευζήν των ζώων. Ο Κάντε έλεγε ότι η βία ε, κατά ενός ζώου είναι βία κατά του ίδιου του ανθρώπου. Θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους για την τύχη των αγκάλκους με εκστατείες σε χάρη στους οργανισμούς που αγωνίζονται γι' αυτό ούτως ώστε να εφαρμοστούν και τα ψηφίσματα για την προστασία αυτών των που έχει ήδη εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη βαρβαρότητα. Ευχαριστούμε Κόρβιν Μίκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιους μήνες πριν είχα πει εδώ σε τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια ότι ο κύριος Σούλτς είναι κάποιος που είναι υπεύθυνο για τις επιτυχίες του εθνικού μετόπου Front στη Γαλλία. Κάποιοι γελιοποίησαν αυτή την τοποθέτηση, όμως από πλευράς Υπουργού Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρθηκε ότι ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιτυχίες του εθνικισμού στην Ευρώπη. Αληθεύει αυτό. Δυστυχώς δεν διδάσκονται το ότι οι αρχές του ότι κάθε δράση προκαλεί μια αντίδραση και σε μονόδρομο όταν κινούμεθα σε ένα μονόδρομο τότε είναι μονόδρομη και η απάντηση που έχουμε. Δηλαδή καταστρέφεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω μία ανακοίνωση να κάνω. Ο κ. Ζανλούκα Μπονάνο, μέλος του Κοινοβουλίου, υπέβαλε έτοιμα στον Πρόεδρο για υπεράσπιση της ασυλίας του στα πλαίσια ποινικών διώξεων από το δικαστήριο του Μπολζάνο.